How are we doing? Okay. While we are trying to connect... Ναι, αφού περιμένουμε με τον κύριο Εμμανουέλ Ντομερόντ που είναι ο διοικητής του πάρκου αυτού να σας υπενθυμίσω ένα πολύ θλιβερό γεγονό που συνέβη πριν από δύο εβδομάδες στο ανατολικό τμήμα της ε, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε θέσει αυτό το θέμα στη μέση διάταξη. Υπήρξε μια επίθεση στο Βιρούγκα, στους Φρουρούς. Έγινε σε 9 Απριλίου, στο Βόρειο Κιβού, στο ανατολικό τμήμα της ε, λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό. Όπως ξέρετε, το Βόρειο Κιβού αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας. Πέντε φρουροί δολοφονήθηκαν και ένας οδηγός. Ένας φρουρούς ε, επέζησε και ε, είναι στο νοσοκομείο. Η επίθεση από την ε, πολιτοφυλακή ΜΑΕΜΑ ήταν η χειρότερη τα τελευταία χρόνια στο προσωπικό του Βιρούγκα και με αυτή την επίθεση ο συνολικός αριθμός των φρουρών που έχουν δολοφονηθεί ανέρχεται σε 175. Αυτοί που δολοφονήθησαν ήταν νέοι μεταξύ 22 και 30. Πριν από 4 χρόνια ο διοικητή του πάρκου, ο πρίγκιπας Εμμανουέλ Ντομερόντα, με τον οποίο επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε τώρα, Τραυματίστηκε ο ίδιος σοβαρά από τρεις ενόπλους. Τα θλιβερά αυτά νέα εξηγούν γιατί ο πρίγκιπς Ντομερόντ δεν είναι εδώ. Ορισμένοι τον είδαμε στο, στην Ολομέλεια του Στρασβούργου της ισομερούς ε, συνέλευσης ΑΚΕΟΚ το 2014. Θα συνομιλήσουμε μέσω της μαγείας ε, της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Εάν οι εμπειρογνώμονές μας ε, καταφέρουν να μας συνδέσουν. Τον έχετε? Λοιπόν, πρώτα θα σας δείξω ένα μικρό βίντεο και μετά θα σας μιλήσει ο πρίγκιψης. j'ai décidé à être gardé par Keka, j'avais 12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 τέτοια μασάκρα. Luogo Dume na Mandike Presque. Kabakia Mukunda. Kabakia mwele familia mwenye alikuwa chunga Le parc a, a beaucoup de, des ennemis.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 Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή μας με βάση την απόφαση του Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου 2015 για την προστασία του πάρκου αυτού ήδη είχε τονίσει ότι οι ένοπλες συγκρούσεις με αντάρτικες ομάδες όπως η ΜΑΙ-ΜΑΙ και η FDLR έχουν κάνει σοβαρέ παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τρομερή βία στο πάρκο αυτό που είναι το, πιο, ε, το κέντρο τη μεγαλύτερη βιοπικιλότητας στην Αφρική και είναι χώρο πολιτιστική προστασία τη UNESCO που περιέχει πολλά εμβληματικά ζώα όπω οι ορεινοί γορίλες, τα οκάπη, οι ελέφαντες και άλλα σπάνια ζώα. Επίση τονίσαμε τότε ότι η εκμετάλλευση και η, η εξερεύνηση για πετρέλαιο στο πάρκο αυτό είναι απόλυτα ασυμβίβαστες, ασύμβατες με την ε, διατήρηση αυτού του πάρκου και του καθεστώτος του ως ε, χώρου της ε, παγκόσμιας κληρονομιάς. Μαζί με τον Μπρίκη Παντεμπερόντα έχουμε εδώ παρόν και τον κύριο Φρανσουά Ξαδιέ Ντουντονέα που είναι υφυπουργό στο Βέλγιο και ε, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Βιρούγκα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντουντονεά που αποδεχθήκατε την, την πρόσκλησή μας. Δεν ξέρω τώρα εάν ε, μπορούμε να συνδεθούμε με τον πρίγκιπα Μερόντ. Μπορούμε Μια συμμετάσχει στη συζήτησή μας. a message after the beep. Is it all right? Is he? Ah. με Timorod, can you hear us? Ε, κύριε πρίγκιπα, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Άριστα. Είμαι εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Σας παρακολουθούμε με τον κύριο Υφυπουργό και μέλος του Διοικητικού σας Συμβουλίου, τον κύριο Ντουντονέα. Σας βλέπουμε. Και είδαμε και ένα σύντομο βίντεο για το πάρκο και παρουσίασα το θέμα των θλιβερών γεγονότων που οδήγησαν το θάνατο 175 νέων και μετά μάλιστα την πρόσφατη επίθεση στον πάρκο. Και πριν από μερικά χρόνια και εσείς τραυματιστήκατε. Ανησυχούμε λοιπόν ιδιαίτερα για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια του προσωπικού και όλων των άλλων μελών του προσωπικού εθελοντών κλπ. που δουλεύουν μαζί σας για το πάρκο. Μήπως σας θέλετε να κάνετε μια σύντομη παρουσίαση και μετά θα καλέσω και τον κύριο Υφυπουργό να μας μιλήσει. Και μετά ε, τα μέλη της Επιτροπής μας θα μπορέσουν να κάνουν ερωτήσεις. Παρακαλώ, πριν και εγώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι παρόν. Σας ευχαριστώ εκ μέρους των αρχών του πάρκου. Και ιδιαίτερα από πλευράς των ε, φυλάκων μας. Και νομίζω ότι um.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 While, while we try and get in back in conversation with Emmanuel de Moreau. Λοιπόν, τώρα τον χάσαμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε τα αίτια αυτών των συγκρούσεων που έχουν προκαλέσει τόσα δεινά 6 εκατομμύρια πρόσφυγες διασκοπισμένοι στο Ανατολικό Κονγκό και δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη που συμβαίνει αυτό έχει ξανασυμβεί ορισμένοι ήμασταν εδώ και παλιότερα έχουν επανειλημμένα σημειωθεί τέτοια πράγματα. Έχει υπάρξει η διαδικασία Κίμπελη, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και όλες οι άλλες ε, ρυθμίσεις για να προστατεύσουμε τα ορυκτά ή διαμάντια από περιοχές σειράξεων. Όμως ε, ορισμένοι με τρομερή επιρροή και τεράστια οικονομική ισχύ χρηματοδοτούν ε, τη δημιουργία ιδιωτικών στρατών και προκαλούν εντάσεις μεταξύ διαφορετικών φυλών για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν ε, αυτές τις ε, πηγές πλούτου. Αυτό είναι ένα διεθνές πρόβλημα που ανησυχεί βέβαια και το κοινοβούλιο μας που δεν έχει στρατό αλλά ανησυχεί και τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να αντιμετωπίσει και άλλη μια προσφυγική κρίση. Βεβαίως έχουμε προσφυγική κρίση στην Συρία και την Τουρκία. Αλλά στην περίπτωση της Αφρικής μόνο λίγες χώρες, ε, το Βέλγιο και ίσω η Γαλλία ασχολούνται με το θέμα αυτό. Οι άλλες χώρες της Ένωσης δεν μοιάζουν να πολύ ενδιαφέρονται εάν οι μαύροι σκοτώνουν Εγώ όμως ανησυχώ και νομίζω ότι και οι Βέλγοι ανησυχούν. Και καλό τον κύριο Υφυπουργό να πάρει το λόγο μέχρι να καταφέρουμε να ξανασυνδεθούμε με τον κύριο, με τον πρίγκιπα Εμμανουέλ του Ευχαριστώ ε, που με καλέσατε. Μου υπενθυμίζει την εποχή που ήμουν και εγώ μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από πολλά χρόνια. Ο κυριότερος λόγος για τα προβλήματα που έχουμε σε πολλές περιοχές της Αφρικής και ιδιαίτερα στο Εθνικό Πάρκο Βιρούγκα είναι η φτώχεια των πληθυσμών της περιοχής. Ένα μεγάλο πρόβλημα στη Βιρούγκα είναι ότι υπάρχουν 4 εκατομμύρια άτομα ζουν σε λιγότερο από ένα εκατομμύριο ε, λιγότερο από μία μέρα περπάτημα από την περιοχή. Και βεβαίως και το κράτος ε, έχει διαχειριστεί από την ανεξαρτησία και μετά άσχημα το πάρκο διάφορες ένοπλες ομάδες εύκολα βρίσκουν ανέργους για να στρατολογήσουν παρά να κάθονται να καλλιεργούν ε, τη λίγη γη της οικογένειάς τους που δεν τους αποφέρει τίποτα. Στο πάρκο Βιρούγκα τι μπορούν να βρουν αυτές οι ένοπλες ομάδες. Αλλά να δώσω το λόγο στον ε, Εμμάνιουελ για άλλη μια φορά.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 Αλλά τι άλλο θα θέλατε να κάνουμε. Ευχαριστώ που αναγνωρίσατε την προσφορά μας. Αλλά είναι σαφές ότι δεν έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Και δεν είναι και οι προοπτικές για το μέλλον πολύ καλές. Απλώς κρατιόμαστε. Το υδροελεκτρικό πρόγραμμα θα μπορούσε να λάβει περισσότερη στήριξη. αν μας πείτε τι θα μπορούσατε να κάνετε για να αυξήσετε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ε, κατασκευής ε, και άλλων σταθμών παραγωγής. Κάτι άλλο. Ε, Α, εδώ είστε, με ακούτε? Όχι πολύ καλά. Right. Do you... Λοιπόν, θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να φτιάξετε και άλλες μικρές ε, μονάδες υδροηλεκτρικής ενέργειας στο πάρκο για να παραγάγετε και άλλο ηλεκτρισμό. Δεύτερον, είπατε ότι τα κέρδη, τα παράνομα κέρδη από ε, τα καμένα δέντρα ανέρχονται σε 100 εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν τίποτα γεωστατικοί δορυφόροι πάνω από το πάρκο που να παρακολουθούν τι συμβαίνει. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να εγκαταστήσουμε κάποιους τέτοιους δορυφόρους. Εύκολο είναι να τους θέσουμε σε τροχιά. Λοιπόν, και επίσης είπατε ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους στην περιοχή, για τους κατοίκους περιοχής. Τι μπορούμε να κάνουμε για να υπάρχουν περισσότερες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 για την ιδιωτική χρηματοδότηση της ανάπτυξης μέσω επιδοτήσεων που συνδυάζονται με ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις. Έτσι, 4 δισεκατομμύρια αναπτυξιακής βοήθειας ε, ήταν η βάση για 70 δισεκατομμύρια ιδιωτικών επενδύσεων. Δημιουργούμε έτσι έναν ενάρετο κύκλο. Υποτίθεται πώ είναι το σχέδιο Juncker, αλλά είναι πρωτοβουλία στην πραγματικότητα της Επιτροπή Ανάπτυξης. Μπορούν να σας βοηθήσουν. Μπορείτε να χρηματοδοτήσετε πολύ περισσότερα προγράμματα από το Ταμείο αυτό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή για να σε ενημερώσουμε για τις δυνατότητες πρόσβασης σε αυτή τη χρηματοδότηση. Καλωσορίζω, όπως έλεγα και προηγουμένως, τον Υπουργό κύριο Φρανσουά Ξαβιέ Ντουντονέα που υποθέτω γνωρίζετε πολύ καλά. Κύριε Υπουργέ, θα θέλετε να πάρετε τον λόγο. Να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Εμμανουέλ Ντομερόντ. Ο μόνος τρόπος για να σωθούν ε, τα εθνικά πάρκα στην Αφρική, μεγάλες περιοχές φύσης, είναι να αναπτυχθεί η περιοχή αυτή να αναπτυχθούν οι περιοχές, οι περιοχές αυτές. Βεβαίως θα χρειάζεται η παρουσία των σωμάτων ασφαλείας για να αντιμετωπιστεί η λαθροθυρία και η παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Αλλά σίγουρα η μεγαλύτερη απειλή για τα εθνικά πάρκα και για τη φύση στην Αφρική είναι η δημογραφική πίεση. Και 70% του πληθυσμού, όπως είπε και ο Εμμανουέλ, είναι άνεργοι. Κάτι άλλο που περιπλέκει την κατάσταση στην περιοχή του πάρκου Βιρούγκα, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Εμμανουέλ, είναι ότι υπάρχει συνεργασία αυτών των ενόπλων ομάδων με τοπικές αρχές. Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να τις εξαλείψει. Τις αντιμετωπίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να τις εξαλείψουμε. Όσο έχουν ισχυρούς ε, δεσμούς αυτές οι ένοπλες ομάδες με τους ντόπιου πολιτικούς, με τους πολιτικούς επιτόπου και πολλές φορές και με τους ε, πολιτικούς σε εθνικό επίπεδο, η Μινούσκο δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά δεν έχει και διάθεση. Οπότε οι φύλακές μας ε, είναι μόνοι στην καταπολέμηση αυτών των ομάδων, αλλά δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Πρέπει να συμμετάσχουν και οι επενδύσεις για να βοηθήσουν τον πληθυσμό και να συνεχιστεί και η μάχη κατά των πιο επιθετικών ενεργειών αυτών των ενόπλων ομάδων στις περιοχές ε, του πάρκου ή γύρω από το πάρκο. Ευχαριστώ. Ε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγιο. Έχουμε τους συνομιλητές μας, έναν εδώ και έναν μέσω του Skype. Παρακαλώ, έχετε Η κυρία Χάουταλα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Υψηλότατε, με ακούτε, ακούτε τη φωνή μου. Σας ακούω. Κοιτάξτε, πρώτα να σας εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τα πρόσφατα θύματα μεταξύ των θηροφυλάκων, τους πέντε αυτούς ε, νέους και τον οδηγό. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, στην Επιτροπή Αναπτύξεως, οφείλουμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη αυτή με κάθε λεπτομέρεια και να συμβάλλουμε όσο μπορούμε στην προσπάθειά σας και χαίρομαι που η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεργάζεται μαζί σας και έχουμε και την ευκαιρία να ρωτήσουμε και τους εκπροσώπους της τι ακριβώς κάνουν τώρα για να ενισχύσουν τη διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Βιρούγκα. Να σας ευχαριστήσω πρώτα για την ε, πολύ ξεκάθαρη και εύγλωτη ε, παρουσίαση των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε στο Πάρκο Βιρούγκα με την έλλειψη κράτους δικαίου, με την έλλειψη στέρεων θεσμών, με το πρόβλημα της ε, ανύπαρκτης απασχόλησης και από το σχέδιο εκθέσεώ μου που θα υποβάλλω μου φαίνεται μάλιστα τώρα σε μισή ώρα σχετικά με την διαχείριση των δασοκομικών πόρων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Σε αυτό δηλαδή με βοηθείτε, μαθαίνω πολλά από αυτά που εξηγείτε και την κατάστασή σας για το ποια πράγματα μπορώ να περιλάβω στην έκθεσή μου. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. εξηγείται εξηγείτε πώς μπορούν να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη γύρω από ε, πάρκα ε, διατήρησης της φύσης. Αν μου επιτρέπετε να ερωτήσω με τη σειρά μου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς βλέπουν την κατάσταση και τις δυνατότητες που έχουν να βοηθήσουν εσάς στο σημαντικό έργο που κάνετε στο Κόγκο. Who speaking on behalf of the Ποιο θα μιλήσει εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, είμαστε δύο εδώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Η Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ, λέγομαι Ντιμάρο. Σα ευχαριστώ για την ε, ερώτησή σα και από τη δική μα ε, σκοπιά, βέβαια, εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μα για τι πρόσφατε απώλειε. Παρακολουθούμε την κατάσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπω είπε ήδη ο πρίγκιπ Τεμερόντ, ε, στηρίζουμε το Εθνικό Πάρκο Βιρόνικα και όχι μόνο για εδώ και τρει δεκαετίε με ε, υψηλό επίπεδο δέσμευση και μακροπρόθεσμη. Ε, είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να επιληθεί βέβαια γρήγορα. Διαθέτουμε πόρους για την υπόθεση αυτή εδώ και πολύ καιρό και θα πρέπει να τεθεί το θέμα και στο ε, προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο. Με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτύξεως έχουμε εγκρίνει ένα πρόγραμμα για το Κονγκό 130 εκατομμύρια ευρώ για να υποστηρίξουμε πέντε εθνικά πάρκα, ορισμένα από αυτά που έχει υποστηρίξει και η UNESCO και τα έχει περιλάβει στην ε, λίστα της Παγκόσμιας Κληρονομιάς Ανθρωπότητας. Χρειάζεται μια ε, ε, συνολική προσέγγιση, δηλαδή και διατήρηση της φύσης και βιώσιμη γεωργία και παραγωγή ενέργειας. Για να σας δώσω μια ιδέα της αναλογίας, είναι 30% διατήρηση και 70% ανάπτυξη και γεωργία και ανάπτυξη γεωργίας. Γιατί λόγω των δημογραφικών πιέσεων, λόγω του πληθυσμού που ζει γύρω από τα πάρκα, αν δεν μπορέσουμε να αφαιρέσουμε την πίεση αυτή από το πάρκο, δίνοντας άλλες δυνατότητες, οικονομικές δυνατότητες, δουλειές στον κόσμο που ζει γύρω από το πάρκο, δεν θα μπορέσουμε να το σώσουμε στο τέλος. αυτά λοιπόν κάνουμε λίγο πολύ. Πρόκειται για μια, όπως είπα, ενιαία προσέγγιση μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Δίνουμε στήριξη και στους θηροφύλακες και στην, για την εκπαίδευσή τους που είναι πολύ σημαντικά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση. Διότι όπως λέχθηκε προηγουμένως η διαχείριση του πάρκου είναι και η μόνη που υπάρχει. Είναι το μόνο ας πούμε κράτος δικαίου που υπάρχει στην περιοχή αυτή. Έχουν και κάποιες ε, εντό εισαγωγών δικαστικέ εξουσίε τι οποίε ασκούν ε, στη βάση των κανόνων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ε, ε, ε, αξιοπρεπούς αντιμετώπισης των συλληφθέντων όσων συλλαμβάνουν εκεί δηλαδή, και ο, η προσπάθεια που κάνουν έχει πάρα πολύ στενή ε, σχέση και με την διατήρηση της τάξης. Σας ευχαριστώ οι άλλοι εκπρόσωποι της Επιτροπής. Δουλεύουμε στη βάση των διαφόρων μηχανισμών που διαθέτουμε. Όπως είπε η Φραντσέσκα έχουμε το 10ο EDF και έχουμε και κονδύλια για το περιβάλλον, τα οποία κινητοποιούμε και προ δύο εβδομάδων κινητοποίησαμε νέο πρόγραμμα για ξυλία που προέρχεται από περιοχή συγκρούσεων στο νότιο μέρος του πάρκου για να επιτρέψουμε στο πάρκο να φτιάξει μια δύναμη άμεση αντίδραση από θηροφυλακέ, αλλά και να προωθήσουμε και τον οικολογικό τουρισμό. Αφενό λοιπόν διαχείριση και ασφάλεια. Από την άλλη μεριά συνεργαζόμαστε με τον Εμμανουέλ Ντεμερότ και την ομάδα του για να προσφέρουμε δυνατότητε επιλογής σε, ε, στους τοπικούς πληθυσμούς και την ομάδα Βερονγκά που ασχολείται και με την λίμνη. Η επίθεση που υπέστησαν όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε θηροφύλακες και ο οδηγός του οχήματος ε, είναι πολύ βαρύ, αλλά ε, παρόλα αυτά κάνουμε μια προσπάθεια να ενισχύσουμε τον οικολογικό τουρισμό για να δείξουμε ότι η πράσινη οικονομία είναι, δίνει μια δυνατότητα για οικονομική ανάπτυξη σε τέτοιες περιοχές και να προσφέρουμε στους νέους οι οποίοι προσελκύονται από τις ντόπιες πολιτοφυλακές και κάποια αξιοπρεπή δυνατότητα επιλογής. Και για το EIP θα, έχουμε την επόμενη, θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα αποστολή μονάδων ενέργειας, σε μονάδες ενέργειας μάλλον. Οι άνθρωποι μας θα πάνε εκεί για να συζητήσουν με τον Εμμανουήλ και την ομάδα του τη δυνατότητα να δοθούν δάνεια για την ανάπτυξη της υδροελεκτική ενέργειας γύρω από το πάρκο και να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε και εγγυήσει ε, της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων για το πάρκο. Και οι συνάδελφοί μου των χρηματοδοτικών μηχανισμών ενδιαφέρονται πολύ να δουν εάν μπορούν να κινητοποιήσουν τις εγγυήσεις αυτές υπέρ του συγκεκριμένου προγράμματος. Και ολόκληρη η διαχείριση ΔΕΦΚΟ συμμετέχει. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτές. Πρόεδρος Ντέβα, ευχαριστώ πολύ. Ντεύκο, από την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Είναι κάποιο παρόν, ναι. Να έχετε να πείτε και εσεί κάτι. Όχι, δεν έχω πολλά να προσθέσω στα όσα είπαν οι συνάδελφοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμμετέχουμε απολύτω. γνωρίζουμε τη σημασία της διασύνδεσης ασφάλειας και ανάπτυξης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για το θέμα αυτό, αυτό είναι κάτι το οποίο ε, ε, είναι πάρα πολύ γνωστό στην ίδια τη λαοκρατική δημοκρατία του Κονγκό και καμιά φορά είναι πάρα πολύ πυκνή η συνολική πολιτική εικόνα και δυσδιάκριτη, αλλά ε, έχουμε την στήριξη των αρχών για το διαθωτικό έργο που κάνουμε για να συνδέσουμε ασφάλεια, ανάπτυξη και προστασία της βιοπικιλίας. Πρόεδρος Ντέβα. Ε, έθεσα και το θέμα των δορυφόρων προηγουμένως. Τι γίνεται, αν θέλετε να παρακολουθείτε την παράνομη δασοκομεία, αυτό είναι προφανές. Γίνεται κάτι τέτοιο, έχετε την ικανότητα να προβλέψετε κάτι τέτοιο. Ερώτηση προς... Ε, Α, εσείς παρακαλώ ορίστε. Ναι, μπορώ να απαντήσω διότι πράγματι μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Κοπέρνικος ζητήσαμε από άλλες υπηρεσίες ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να φτιάξουν ένα σύστημα παρακολούθησης προστατευόμενων περιοχών στην Αφρική. Προ λίγων μηνών έγινε και αποστολή του Κοινού Κέντρου Ερευνών που αναλύει τις εικόνες αυτές, τις φωτογραφίες αυτές για να διαπιστώσουμε την έκταση της παράνομης ε, υλοτομίας στην περιοχή του Πάρκου Βιρούνκα, όπως κάνουμε και σε άλλα 15 άλλα πάρκα της, ε, της ε, Αφρικής. Είναι, είναι απολύτως δυνατόν αυτό. Έχουμε και ε, ευκρινείς εικόνες σε επίπεδο 10 μέτρων με τους δορυφόρους που διαθέτουμε. Έχουμε λοιπόν εικόνες στην, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών ε, υψηλότατε θέλετε να πείτε κάτι σχετικά. Μπορείτε να συνομιλήσετε με τον εκπρόσωπο που μόλις μίλησε για τα θέματα αυτά. Ενδεχομένω να μπορείτε να δείτε και ποιος, ε, ποιοι είναι οι επιτιθέμενοι σε περιπτώσεις ε, επιθέσεων. Άλλος κανείς, παρακαλώ και των συναδέλφων. Ορίστε εσείς κύριε Βένταν. Απλή ερώτηση διότι προ μια ώρα κάναμε συζήτηση εδώ για τις μεταρρυθμίσεις για την Αφρικανική Ένωση. Ε, προτάσεις για το θαυμάσιο αυτό τρόπο, τόπο όπου ωστόσο χάνονται ανθρώπινες ζωές στην προσπάθεια διατήρησης της ε, φυσικής ομορφιάς. Το ερώτημα είναι ποια είναι η θέση της Αφρικανικής Ένωσης για τα πράγματα. Για παράδειγμα, η σταθεροποίηση κατάσταση στο Κονγκό σε σχέση και με τις ε, νέες εκλογές. Ίσως και εκεί μπορούν να ληφθούν κάποιες πρωτοβουλίες, διότι το πάρκο Βιρούνγκα δεν βρίσκεται μόνο στην επικράτεια του Κονγκό, ε, καλύπτει επικράτειες και άλλων χωρών. Ποια είναι η θέση της Αφρικανικής Ένωσης ε, εν προκειμένου. Ορίστε, ευχαριστώ. Yes, from the years. Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ευρύτερο πολιτικό θέμα αυτό βεβαίω που θίγεται εδώ. Είναι προφανέ ότι από, εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργαζόμαστε στενά με του συναδέλφου μα τη Αφρικανική Ένωση. Ο πρόεδρο τη Επιτροπή Αφρικανική Ένωση, κ. Μουσαφάκη, επισκέφθηκε δύο φορές του τελευταίους μήνες ε, την χώρα αυτή και είναι σε άμεση επαφή με τον ίδιο τον πρόεδρο και έχει εξηγήσει πολύ καθαρά την θέση της Αφρικανικής Ένωσης και έχει ενισχύσει, έχει, έχει προσφέρει ε, στήριξη στην, ε, ε, στις φωνές που ζητούν εκλογές. Υπάρχει λοιπόν σημαντική στήριξη από πλευράς της Αφρικανικής Ένωσης, με την οποία, όπως είπα, συνεργαζόμαστε στενά. Και έχοντας την έδρα μου στην Κινσάσα, ε, συναντώμε με τον συνάδελφο της Αφρικανικής Ένωσης τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Είναι λοιπόν ευρύτατη η συμφωνία μας, μεταξύ μας συνένεση σχετικά με το ότι είναι αναγκαίες εκλογές. Και αυτό στηρίζεται και από την Αφρικανική Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους διεθνείς φορείς στην Κινσάσα και βεβαίω και άλλους που ενδιαφέρονται για την κατάσταση στην ε, λαοκρατική δημοκρατία του Κονγκό. Ευχαριστώ πολύ, Ντέβα. Με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι καθόμαστε όλοι εδώ ανταλλάσσοντας ε, απόψεις στη βάση, ε, μάλλον με τη βοήθεια μιας πολύ σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει και να προστατευτούν κάποιοι ε, άνθρωποι που το αξίζουν. Άλλος επιθυμεί κανεί. Ωραία, μου φάνηκε θαυμάσια η συζήτηση αυτή. Ποιο είναι το επόμενο βήμα. Η Επιτροπή έχει κάτι να προτείνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το Εθνικό Πάρκο Βιρούγκα. Έχουμε μάλιστα σχέδια να εντείνουμε την υποστήριξη αυτή και για τον τομέα παραγωγής ενέργειας και για τον αγροτικό τομέα με τα κονδύλια του 11ου ε, Ευρωπαϊκού Ταμείου Αναπτύξεως, πράγματα τα οποία βέβαια πρέπει να συζητήσουμε με τους ε, ομολόγους και συνομιλητές μας, το ε, Εθνικό Ινστιτούτο του Κονγκό για την προστασία της φύσης, ε, με το οποίο συνεργαζόμαστε καλά και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να αυξήσουμε την υποστήριξη. Και χρησιμοποιούμε όλου του μηχανισμούς που διαθέτουμε με συντονισμένο τρόπο. Αυτή άλλωστε είναι και η δέσμευσή μα απέναντί σα. Η ΕΤΕΡΑ εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Δεν είναι μόνο χρηματοδοτική η υποστήριξη που χρειάζεται, το πάρκο Βερόνικα χρειάζεται και ορατότητα. Να, ε, να φαίνεται καθαρά τι είναι, που βρίσκεται κλπ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό επίση. Κάτι που νομίζω δεν είπε ο Εμμανουέλ Ντεμερόντ είναι ότι το πάρκο έχει προταθεί από τον Αρχιεπίσκοπο Τούτου για βράβευση με βραβείο Νομπέλ. Να ένας τρόπος που μπορούμε να καταστήσουμε πιο ορατό στα μάτια της διεθνούς κοινή νόμης αυτήν την περιοχή. Και εκεί επίσης θα χρειαστούμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διασφαλίσουμε ώστε θα παραμείνει ε, κάτω από τα μάτια της διεθνούς το ε, πάρκο αυτό. Ο πρόεδρος Ντέβα. Μήπως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διορίσει, να ορίσει κάποιους ειδικού εκπροσώπους ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει στο Εθνικό Πάρκο. Εμμανουέλ, ε, εσείς βρίσκεστε εκεί επί τόπου, ενώ εμείς είμαστε εδώ. Ε, κάπως μακριά. Πώς, πότε θα θέλατε να επανέλθουμε. Ε, κάπως μας προσφέρατε μια πρόκληση και θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Σας ρωτώ λοιπόν να μας πείτε εμάς πότε θέλετε να επανέλθουμε καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις. <laughs>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 um, from our viewpoint on the ground, um, that you know we could reach a turning point um, with a a, a more positive um, light at the end of the tunnel. Thank you. um, Colleagues, ladies and gentlemen, I want to thank... Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια που, τις προσπάθειες που καταβάλλετε όλοι για το θέμα αυτό. Και ε, συγχαίρω τι εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι θαυμάσιε απαντήσει που έδωσαν. Και για εσά που ήρθατε από την Κινσάσα για να ε, τη στη συζήτηση σας, ε, εύχομαι καλή τύχη, Εμμανουέλ, και θα παραμείνουμε σε επαφή. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Υπουργό που ε, προσήλθε εδώ και μιλώ για κάτι το οποίο είναι δυνατόν να γίνει. Κάτι το οποίο, στο οποίο μπορούμε να συμβάλλουμε στις προσπάθειές μας για να επιφέρουμε κάποιες αλλαγές. Και νομίζω ότι θα αποτελέσει και μια καλή δοκιμασία για όλους και όλους μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και πάλι. Συνεχίζει ο πρόεδρος για τα δασοκομικά τώρα που είναι το επόμενο θέμα. Έχουμε Ε, πρέπει να δούμε, συνεχίζει ο πρόεδρος το θέμα λογοδοσία και διαφάνεια στην διαχείριση φυσικών πόρων σε αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίω για πόρους δασών. Που αυτό, ξαναλέω, είναι το αντικείμενο του, της επόμενης συζήτησης που χειρίζεται η ικανή συνάδελφός μας Χάιντι Χάουταλα, που είναι και συγγήτρια για το θέμα αυτό. Και θυμάστε ότι στην προηγούμενη συνάντηση κάναμε μια πρώτη συζήτηση με παρουσίαση και του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και με παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους, τις βασικές αιτίες της ε, αποψήλωσης δασών που και οι κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται ποιες είναι οι αιτίες αυτές και στην τελευταία συνάντηση επαναλάμβαμε την ανάγκη να υπάρξει υπεύθυνη διαχείριση των δασών. Και σήμερα θα γίνει συζήτηση στη βάση του σχεδίου ψηφίσματος που έχει επεξεργαστεί η κυρία Χάουταλα. Και ας αρχίσουμε με την δική της πρώτη τοποθέτηση. Σα ευχαριστώ. Δεν μπορώ να κατηγορήσω όσου έφυγαν, ε. αλλά λυπούμε γιατί είναι άμεση η συσχέτιση της προηγούμενης συζήτηση με το σχέδιο έκθεση. Τουλάχιστον όμω δύο συνάδελφοι παραμένουν στην αίθουσα, αν δεν κάνω λάθος, και με ευγνώμονα σε αυτούς τους δύο. Έχουμε μια είχαμε μια μελέτη, είχαμε μια ακρόαση για τον τίτλο αυτής της ε, έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας για τη διαφάνη διαχείριση ε, των πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες η υπόθεση των δασών. Έχει δοθεί ας πούμε, περισσότερη προσοχή στην εξόριξη και τους ορυκτούς πόρους και εκεί ε, υποστηρίζουμε την ε, διαφάνεια και τη λογοδοσία στη χρήση του σε σύγκριση με άλλους πόρους όπως τα δάση που είναι επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι των ανανεώσιμων πόρων αλλά και της φύσης ε, του πλανήτη. Εγώ έχω συνεργαστεί στενά με τους δύο άλλους συντάκτες γιατί η Επιτροπή Περιβάλλοντος σωστά διεκδίκησε κοινή αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για αρκετά τμήματα που ελπίζω θα συνδεθούν με τη δική μου δουλειά που γίνεται από την οπτική της ανάπτυξης. Και υπήρξε και μια εξαιρετική γνωμοδότηση στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου που προσθέτει μια ακόμα διάσταση στην έκθεση αυτή. Ήταν μια μοναδική εμπειρία γιατί μπόρεσα, μπόρεσα να συνεργαστώ με δύο άλλους ηγητές και διαπιστώσαμε ότι ο καθένας μας είχε μια διαφορετική εικόνα, μια διαφορετική μάλλον οπτική για το θέμα της διαχείρισης των δασών. Συμπίπτει δε αυτό με την ε, δημόσια, αρκετά δημόσια συζήτηση ή ε, τουλάχιστον δημόσια για όσους προσέχουν την ανάπτυξη και την ε, δασοκόμια. Με συγχωρείτε, αλλά ε, έχει πάρα πολύ φασαρία. Μπορείτε να βγείτε από την αίθουσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα δράση για την αποψήλωση των δασών και την υποβάθμιση των δασών από πλευρά Ένωση. Ε, ένα από του βασικού έξονε τη πρότασή μου είναι ότι θα πρέπει να καλέσουμε την Κομισιόν να ξεκινήσει άμεσα μια ε, περιστατωμένη μελέτη αξιολόγησης για να μπορέσουμε να συστήσουμε ένα τέτοιο πλάνο για την αποψήλωση των δασών και την υποβάθμιση των δασών και συγκεκριμένα ρυθμιστικά μέτρα ώστε καμία αλυσίδα παροχής ε, η αλυσίδα που χρηματοδοτείται από την Ένωση να μην προκαλούν την αποψήλωση των δασών. Και έρχομαι στο κεντρικό θέμα που πρέπει να δούμε εδώ και είναι βέβαια η Ατζέντα 2030. Ναι, Διάφοροι βιώσιμοι στόχοι συνδέονται με την δασοκομεία και τη διαχείριση των δασών και συγχαίρω τον Εμμανουέλ Τεμερότ που πραγματικά εξηγεί περί τίνος πρόκειται από το κράτος δικαίου μέχρι τη δημιουργία βιώσιμων ε, θέσεων απασχόλησης στην καταπολέμηση του εγκλήματος και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πολύ πιεστικές ε, ε, προκλήσεις όσον αφορά την απώλεια βιοπικιλότητας και βέβαια και η φτώχεια και πρέπει να τονίσουμε ακόμη περισσότερο από ό,τι παλιότερα την συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής να συμβάλλουμε στην πολιτική βιοκαυσίμων ε, και την εμπορική πολιτική μεταξύ άλλων. Αλλά ευτυχώς η Ένωση έχει ήδη στη διαθεσή της σημαντικά μέσα όπως το πρόγραμμα δράσης μπλε και οι εθελοντικές, ε, μάλλον οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης, εθελοντικής εταιρικής σχέσης που εγκρίνονται από, από όλα τα μέρη για να βελτιωθεί η δασοκομεία στην ε, τις χώρες εταίρους. Όμως από μόνο του αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα ότι ο των δασών σε μεγάλο βαθμό προκαλείται από τη γεωργία. Για πολλούς και διάφορους λόγους βέβαια. Ε, και επίσης πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε το θέμα της ξυλίας που προέρχεται από ζώνες ε, εμπόλεμων ε, σειράξεων. Μιλήσαμε για τα ορυκτά από τέτοιου είδους εμπόλεμες περιοχές. Τώρα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη ξυλία από εμπόλεμες περιοχές. Η παράνομη ξυλία είναι μία από τις πέντε μεγαλύτερες πηγές περιβαλλοντικών εγκλημάτων και όλα αυτά έχουν να κάνουν με οικονομίες offshore και την μεταφορά ε, πόρων από εγκληματίες σε σκιώδεις περιοχές, σε νεφελώδεις περιοχές, άγνωστες περιοχές και παραδείσους. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι ε, Ε, έχει να κάνει το θέμα, το πρόβλημα της παράνομης υλοτομίας είναι ε, απόλυτα συνδεδεμένο με το θέμα της κατοχής γης. Ε, θα πρέπει να δούμε, είναι ένας από τους φραγμούς στην αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας. Πώς θα συνδυαθεί η, συντήρηση με την οικονομική ανάπτυξη ή θα, μπορούσαμε να μάθουμε πολλά από το Βιρούγκα. η ε, αποψήλωση των δασών δεν συμβαίνει εν κενό. Ε, η Ένωση έχει στην διάθεσή της διάφορες ε, νομοθεσίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως έμπνευση για να συνταχθεί νομοθεσία για την υλοτομία και μιλώ εδώ για την νομοθεσία περί παράνομης αλληλείας και περιορικτών από ζώνες εμπόλεμων συγκρούσεων. Ο ιδιωτικό τομέα μπορεί να παίξει βασικό ρόλο στην βιώσιμη υλοτομία όμως χρειάζεται σαφή ε, ε, νομοθεσία περί δέουσας επιμέλειας και αυτό ακριβώς δήλωσε και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου στην ψηφοφορία της. Χρειάζεται λοιπόν ξεκάθαρη νομοθεσία περί δέουσας και με χαρά βλέπω ότι επιτέλους η Κομισιόν θα προτείνει μια μελέτη αντικτύπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο Μάλλον, για σχετικά με την νομοθεσία περί δέουσας επιμέλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, Επίση, θα πρέπει να εξετάσουμε λεπτομερώς τη δυνατότητα χρήσης μιας σήμανσης ειδική για προϊόντα που χρησιμοποιούν εγκεκριμένη ξυλία ε, ε, εξάλλου χρησιμοποιούμε πολλούς, ε, απορροφώνται πολλοί πόροι για να χρησιμοποιείται αυτό το σύστημα νομιμότητας της ξυλίας. Γι' αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίζουν και οι καταναλωτές. Έχει εγκριθεί αυτό το σύστημα, χρησιμοποιείται στην Ινδονησία και θέλουμε να χρησιμοποιηθεί συντόμως και στην Γκάνα. Ε, ελπίζω να κάλυψα τις κεντρικές ε, πτυχές ε, της διαφανούς διαχείρισης των δασών και ελπίζω ότι από κοινού θα μπορέσουμε να καλέσουμε την Επιτροπή να κάνει το, τη δουλειά της. Ναι, σας ευχαριστώ. Ο Σεμπ, Dance. Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντα την εισηγήτρια για την εξαιρετική τη εργασία σε αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι εύκολο, όπω είπατε, δεν είναι εύκολο να συνδυαστούν οι διάφορε, τα διάφορα σε πτυχές ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας περί και όντως η εργασία περί των ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ε, παράδειγμα ώστε να μπορέσουμε να συνδέσουμε όλες αυτές τις αλυσίδες. Έχουμε κάνει προσπάθειες απόπειρες στο παρελθόν όπου το θέμα της αλυσίδας προμηθειών έχουν, έχει δημιουργήσει πρόβλημα γιατί ακριβώς δεν υπήρχαν όλες, όλοι οι κρίκοι. Και για την ξυλία θα πρέπει να γίνει το ίδιο. Να ευχαριστήσουμε ε, τους συναδέλφους από τις επιτροπές που γνωμοδότησαν ε, γιατί υπέβαλαν πολύ καλές συστάσεις και θα βρούμε κοινό έδαφος. Αυξανόμενα ε, αναγνωρίζεται ο ρόλος της δασοκομείας, της υλοτομίας και το πώς αυτή μπορεί να συμβάλλει στην ανάσχεση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων βέβαια των δικαιωμάτων γεωκτησίας των αυτοχθόνων πληθυσμών. Βεβαίως ε, ανταποκρινόμαστε στο θέμα της δασοκομείας αλλά και στις δεσμεύσεις του Παρισιού και των ε, στόχων της χιλιετίας. Θα πρέπει η επιμέλεια να επιβληθεί και στην ξυλία όπως έγινε και με τα διαμάντια. Ήδη υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν συγκεκριμένα ε, προγράμματα για την ξυλία. Έχουν γίνει πολύ καλά βήματα σε κάποιες χώρε προς την εφαρμογή αυτών των, ε, προγραμμάτων. Και... Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι. αλλά και να εξασφαλίσουμε ότι το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η γνώση και η τεχνογνωσία που προέρχεται από τους αυτόχθονους πληθυσμούς, αυτόχθονες πληθυσμούς να ε, τεθούν σε εφαρμογή, να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν. Να βρούμε τρόπους να μειώσουμε την υλοτομία και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από την ξυλία και από προϊόντα όπου τα δάση έχουν πλέον εξαλειφθεί. Γι' αυτό και η πιστοποίηση είναι πολύ σημαντική. Ε, έχουν ε, μπορέσει δεν να αποκατασταθούν και ο στόχος είναι μέχρι το 2030 να αποκατασταθούν εκατομμύρια εκατομμυρίων ε, ε, αποψηλωμένων δασών. Όπως είπα, ελπίζω πως θα βρεθεί κοινό έδαφος και συμφωνία από όλο το φάσμα των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ, ο κύριος Ντέβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την Heidi αλλά και την εξαιρετική της έκθεση. Διερωτώ με αν θα... και εσείς μιλάτε για αποψήλωση των δασών και εσείς μιλάτε για αποκατάσταση, αλλά πόσα δάση έχουν ξαναφυτευθεί Δεν έχω ιδέα τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Πόσα εκτάρια το χρόνο, ας πούμε, ξαναφυτεύονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήταν σκόπιμο να ελέγξουμε αν είναι εδώ κάποιος από τους εκπροσώπους της Κομισιόν και αν το γνωρίζει, γιατί εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Υποψιάζομαι πως η αποψήλωση των δασών είναι η τάση και όχι η εκνεοφύτευση. Αλλά φυσικά ε, ε, και όχι αναδάσωση, αλλά ε, αποψήλωση σημαίνει απερίμωση, απώλεια της επικοινότητα, ενώ η αναδάσωση σημαίνει και θέσεις απασχόλησης, παραγωγή, τραφήμων και ένα σωρό άλλες ε, ευνοϊκές εξελίξεις. Ευχαριστώ. Τώρα, ε, συνάδελφοι, η συνάδελφος από την Κομισιόν. Παρακαλώ, ήρθατε. Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω την ε, κυρία Χαουτάλα. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Και εκτιμούμε ιδιαίτερα και τις σκέψεις και τις διατυπώσεις για το πρόγραμμα δράσης, για τα δάση και για την αναγνώριση της εργασίας που έχουμε κάνει. Αναγνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα δράσης βεβαίως δεν αντιμετωπίζει όλα τα θέματα η αποδάσωση συνεχίζεται. Καταστροφή των δασών. Πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όπως είπατε είναι πολύ περίπλοκο, περίπλοκο θέμα με πολλές διακλαδώσεις. Πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικά. Και εκτιμούμε αυτή την έκκληση για μελέτη εντεκτύπου που κάνατε. Πολύ σημαντική. Για να αντιμετωπίσουμε σωστά το θέμα. Και να γίνει ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους. Ως ΔΕΒΚΟΜ θα διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν όλα αυτά. Και αν πρέπει να κάνουμε ήδη ευθύ εξ αρχής μια πιο περιορισμένη διαβούλευση, θα μπορούσε να βοηθήσει την περαιτέρω δουλειά μας από αυτού. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι να μεταφέρουμε τα προβλήματα από τα δάση σε άλλες μορφές χρήσης της γης και οικοσυστήματα. Ένα εκατομμύριο εκτάρια ανά έτος αναδασώνονται, ε, αλλά κυρίως είναι στη Λατινική Αμερική, όχι παγκοσμίω. Πρέπει να το δούμε αυτό. Και ε, δεν θέλουμε αυτά που κάνουμε να έχουν επιπτώσεις σε άλλου τύπου οικοσυστήματα όπως τα λιβάδια. Θέλουμε να δημιουργηθούν ε, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Δεν θέλουμε, για παράδειγμα, οι προσπάθειες για να μην αξιοποιούνται τα δάση να στραφούν κατά γεωργών που σε άλλες περιοχές, ιδιαίτερα στην Αφρική, εργάζονται σε επίπεδο απλώς επιβίωσης ως γεωργοί. Πρέπει λοιπόν από πλευρά ε, συνεργασία για την ανάπτυξη να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώ αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό. Όπω και εσεί πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο τους εξωτερικούς μας εταίρου, αλλά και ε, δικό μας από πλευρά ε, ζήτησης. Πρέπει να συνεχιστούν λοιπόν οι εσωτερικές διαβουλεύσεις με διάφορα άλλα τμήματα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο με τη Γενική Διεύθυνση ΕΝΒΙ αλλά και Γεωργία, Εμπόριο και άλλες γενικές διευθύνσεις που μπορούν να μας δώσουν ε, τα αναγκαία εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με σωστό και βιώσιμο τρόπο. Πρέπει λοιπόν να είναι συνεπής η αναπτυξιακή πολιτική για τέτοια ακριβώς θέματα Μόνο έτσι θα επιτύχουμε. Όταν προτείναμε τον κανονισμό που έχει μεγάλη σημασία για τα θέματα αυτά. Εξετάσαμε εάν στα κράτη-μέλη υπήρχαν εθνικές ρυθμίσεις που θα μας επέτρεπαν να ανοιχνεύσουμε τα προϊόντα παράνομης υλοτόμησης που μπαίνουν στην αγορά και ανακαλύψαμε ότι μόνο η Γαλλία είχε κατάλληλη νομοθεσία που θα επέτρεπε τη δίωξη όσων εμπλέκονται στην παράνομη υλοτόμηση. Θα πρέπει να γίνει κάτι παρόμοιο για οποιοδήποτε κανονισμό που θα θέλουμε να προτείνουμε για τα προϊόντα που προκύπτουν από την ε, καταστροφή των δασών. Γιατί ξέρετε, αλλάζουν οι μορφές ιδιοκτησίας της γης για την καλλιέργεια φινικόδενδρων και κοκοφινίκων για την παραγωγή ελαίου, από, φινικελαίου και ε, ελαίο από καρίδες, καριδελαίο. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το εξωτερικό πρόγραμμα επενδύσεων, τους διάφορους πυλώνες του, για να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε πιο βιώσιμες ιδιωτικές επενδύσεις σε χώρες με τις οποίες συνεργαζόμεθα, που εξάγουν προς την Ένωση. Επίσης πρέπει να μιλήσουμε με τους εταίρους γιατί υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στη ζήτηση. Η Ευρώπη δεν είναι η μόνη περιοχή που καταναλώνει προϊόντα δασών. Πρέπει να συζητήσουμε με την Κίνα και την Ινδία, όπως για παράδειγμα κάνουμε σε άλλους τομείς με την Κίνα, που είναι μια χώρα που ε, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Οι κανόνες ιδιοκτησίας της γης είναι πολύ σημαντικοί και στα πλαίσια του προγράμματός μας για το 2018 θα κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό. Αλλά είναι περιορισμένη αυτή η πρωτοβουλία. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό. Στη συμφωνία που έχουμε με την Ονδούρα έχουμε για πρώτη φορά εισαγάγει την έννοια της ε, εκ των προτέρων ε, ενημερωμένης ε, συνένεσης. Να δούμε αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό για να εμπλέξουμε σωστά τους αυτόχθονες πληθυσμούς, ούτως ώστε να μπορέσουν να συνενέσουν ε, με τα λόγου γνώσεως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Σοντάλ για αυτή την ενημέρωση. Λοιπόν, Άιντι, θες να προσθέσεις τίποτα. Ναι, νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα ε, κατηγορηματική η έκθεσή μας με τις ε, συνεισφορές της ίντα και της ένβη. Ε, Άρα θαυμάσια δουλειά. Για να καταλάβουμε πόσο ευαίσθητα είναι τα θέματα αυτά, θα γνωρίζετε ότι χώρες που παράγουν φινικέλαιο ανησυχούν ιδιαίτερα από τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δεύτερη οδηγία για τις ανανεώσιμες που είναι σε φάση τριμερούς διαλόγου. Ε, κάθε μέρα μου ζητάει η Ινδονησία να συναντηθούμε για να ε, μπορέσουν να επηρεάσουν τον τριμερή διάλογο. Νομίζω ότι θα μπορέσει να βρεθεί λύση που να μην αντιτίθεται στους παγκόσμιους κανόνες για το διεθνές εμπόριο του ΠΟΕ, αλλά αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε μέσω της ανανεώσιμης οδηγίας τα βιοκαύσιμα, έχουμε δικαίωμα να απαιτήσουμε να είναι βιώσιμης προέλευσης. Ελπίζω όλοι αυτοί η τρικυμία εγκρανίου που είναι λίγο μεγαλύτερη τώρα από τρικυμία εγκρανίου μπορεί τελικά να οδηγήσει σε συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι στις χώρες που καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα υπάρχει πραγματική απέτηση για βιωσίμως παραγόμενα δασοκομικά προϊόντα. Και καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μου και χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι αυτές οι εθελούσιες ε, συμφωνίες έχουν αλλάξει την κατάσταση επιτόπου. Άρα μπορούμε να επιτύχουμε αρκετά πράγματα, γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια κλιματική πολιτική. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Χάιντι, που ήμουνα, προθεσμία για τροπολογίες, 15 Μαΐου, 12 το μεσημέρι. Έκλεισε προς το προσωπικό μας. να ενημερώσετε ότι οι τροπολογίες πρέπει να έχουν σχέση με το κείμενο. Όχι εκατοντάδες τροπολογίες που τελικά ε, νερώνουν τόσο πολύ το κείμενο. Ίσως αυτό το κάνουν γιατί ορισμένα site σημειώνουν πόσες τροπολογίες έχει υποβάλει ο κάθε ευρωβουλευτής. Μα δεν είναι ο καλύτερος τρόπος αυτός για να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Η μας καλεί να σκεφτούμε τι πραγματικές επιπτώσεις επιτόπου έχουν οι ενέργειές μας. Να είναι σύντομες και σχετικές οι τροπολογίες. Ίσως οι ομάδες και οι συντονιστές να μπορούν να το αναλάβουν αυτό. Ευχαριστώ πολύ Χαίτη, και θα το συζητήσουμε τον Ιούνιο. Περνάμε στο σημείο 23. Ώρα ρωτήσω. θα το συζητήσουμε πριν το 22. Γιατί το 22 θα το συζητήσουμε μαζί με την Επιτροπή Προϋπολογισμών θα έρθουν στη συνεδρίασή μας σε λίγο. Δύο ερωτήσεις έχουμε για την ώρα ερωτήσεων. Η πρώτη είναι τον Ενρίκε Γκερέρο Σαλόμ. Ιδιαίτερα επίκαιρη. Αφορά τη διάσκεψη για τη Συρία. Πού λαμβάνει η χώρα. Εδώ, στις Βρυξέλλες, σήμερα και αύριο. Ενρίκε, θα διαβάσω την ερώτηση. Ε, να, ε, να ξέρουν οι παρευρισκόμενοι επί περί πρόκειται και θα δώσω λόγο στον Ερή μετά την αντίδραση της Κομισιόν. Είχαν ε, γίνει υποσχέσεις το 2016 και 2017, υποσχέσεις λοιπόν, αλλά μόνο 33% των υποσχέσεων έχουν εκταμιευθεί. Οπότε η ερώτηση. Τι ποσά υποσχέθηκαν, τι έχει δοθεί τι αναμένετε για τη χρηματοδότηση στην επόμενη διάσκεψη. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα απαντήσει την ερώτηση. Ποιο θα απαντήσει από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Υπάρχει κάποιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν είμαι εγώ το μόνο που να σα πω. Συγγνώμη. Εγώ είμαι με την, ε, από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είχαμε συνεργαστεί με την ΤΕΒΚΟ. Θα είναι εδώ σε 5-10 λεπτά. Συγγνώμη για καθυστέρηση. Ωραία, να πω στους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι χρόνοι είναι όλοι δεκτική. Α, στις 5 και 20 θα πάρω το χρόνο. Είναι δεκτική οι χρόνοι γιατί αλλάζει η μεσή Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να έρχεστε μόνο τη συγκεκριμένη στιγμή, πρέπει να έρχεστε λίγο νωρίτερα. Για τη δική μου ερώτηση είναι κανεί. Από την ΤΕΒΚΟ, για τη δική μου ερώτηση. Α, μόλι ήρθατε. Είστε από την ΕΚΟ. Από την ΤΕΒΚΟ είναι κανεί για να απαντήσει τη δική μου ερώτηση. Για την ΑΓΚΟΑ. Λοιπόν, ωραία, κλείνω το μικρόφωνο για να δούμε τι γίνεται. No, no, I, So, Enrique, we're going to wait for your question. Λοιπόν, Enrique, θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο για την ερώτησή σου. Και έχουμε και μία συμπληρωματική ερώτηση, μία περώτηση, ο Νόρμπερτ και εγώ. Άρα πρέπει να είναι παρόντες οι αρμόδιοι για να ακούσουν ε, τις επιπλέον ερωτήσεις μας. Οπότε, η δεύτερη ερώτηση είναι η δική μου ερώτηση. Περί πρόκειται είναι για τα μεταχειρισμένα ρούχα. Μια σειρά από κάτι μέλη της Ανατολικής Αφρικής ήθελαν να σταματήσουν σταδιακά την εισαγωγή μεταχειρισμένων ρούχων γιατί είχε αρνητικές επιπτώσεις στον κλάδο το δικό τους της ένδυσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απείλησαν να, να σταματήσουν την πρόσβαση στην αγορά τους των ε, χωρών που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΑΓΚΟΑ που είναι ο νόμος για την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες για την Αφρική. Οι περισσότερες αφρικανικές χώρες όταν ε, απειλήθηκαν με αυτόν τον τρόπο ε, υποχώρησαν. Αλλά η Ρουάντα όντως απαγόρευσε την εισαγωγή μεταχειρισμένων ρούχων. Και οι Ηνωμένε Πολιτείες ανέστηλαν την πρόσβαση των προϊόντων της Ρουάντα από την αγορά τους. Αλλά από ό,τι κατάλαβα η Ρουάντα δεν έχει τρομερό εμπόριο με τις ΗΠΑ. Αλλά το θέμα είναι γενικότερα τα μεταχειρισμένα ρούχα. Το θέμα είναι εάν έχουμε εμείς κάποιους κανόνες για την αγορά μεταχειρισμένων ρούχων. και αν ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει αυτό το εμπόριο στον κλάδο και στις εσωτερικές αγορές. Γιατί τα προϊόντα ένδυσης, τα κλώστο υφαντουργικά σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες είναι η αρχή της εκβιομηχάνησης. Ανησυχώ δηλαδή ότι κάποιες ε, πλούσιες χώρες για να προστατεύσουν τη δική τους δευτερογενή αγορά ρούχων φύγουν ε, τον κλάδο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είστε από την Digi Inta. Από την DG Trade είστε. Α, DG Trade. Με συγχωρείτε, δεν έχω το όνομά σα, αλλά παρακαλώ, οπότε πείτε μας το όνομά σα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, υπήρξε κάποια παρανόηση. Λέγομαι Θάνος Ράμος. Εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση Trade και ιδιαίτερα για την κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής. Από ό,τι κατάλαβα η κατάσταση έχει ως εξή Και είναι πολύ απλή. Από το 16 και μετά. Οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν έγιναν κατόπιν από διαβούλευση με εμάς ε, οι ενέργειες τελικά δεν έγιναν πραγματικότητα αυτές οι απειλές στις 30 ε, Μαρτίου οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν την κυβέρνηση της Ρουάντα ότι είχαν την πρόθεση να αναστείλουν όλα τα προϊόντα ένδυσης να αναστείλουν δηλαδή την πρόσβαση χωρίς δασμούς στην αγορά των ΗΠΑ όλων των προϊόντων ένδυσης μέσω αγκόα εντός 60 ημερών εάν δεν αλλάξει στάση η Ρουάντα. Άρα δεν έχει υπάρξει εφαρμογή αυτού του μέτρου για να αποτιμήσουμε την, τον αντίκτυπό του. Εάν λοιπόν εφαρμοστεί θα αφορά μόνο ρούχα. Οι εξαγωγές από τη Ρουάντα στις ΗΠΑ τέτοιων προϊόντων είναι πολύ μικρές. Από ό,τι ξέρουμε με βάση τη δική μας ε, πληροφόρηση είναι 5%. Είναι δηλαδή 1,5 εκατομμύριο δολάρια για το 2017. Σε ένα σύνολο εξαγωγών 32,9 εκατομμυρίων από τη Ρουάντα προς τις ΗΠΑ. Τώρα, τι αντίκτυπο θα είχαν αυτά τα μέτρα. Δεν το έχουμε εξετάσει. Γιατί δεν έχει εφαρμοστεί. Αλλά κάποιες μελέτες ε, που υπάρχουν Ενώ η κυβέρνηση της ε, Ρουάντα θεωρεί ότι αν απαγορεύσει αυτή την εισαγωγή μεταχειρισμένων ρούχων ε, θα δημιουργηθούν 25.000 θέσει εργασία. Εμείς δεν είμαστε σίγουροι. Υπάρχει μία μελέτη γενικότερα για την αγορά μεταχειρισμένων ρούχων Αυτή η μελέτη είναι περσινή. Πολύ πρόσφατη και καταλήγει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν εισόδημα από τα μεταχειρισμένα προϊόντα ενώ θα εξακολουθήσουν μεταχειρισμένα ρούχα ενώ θα εξακολουθήσουν να έχουν τα ωφέλη και από την αγκώα και οι χώρες αυτές θα μπορούσαν να έχουν τα ωφέλη και από την αγορά μεταχειρισμένων ρούχων και από την αγκώα ενθαρρύνοντας και τον τομέα της παραγωγής προϊόντων ένδυσης. Η Κένια, η Ουγγάντα και η Τανζανία που επίσης επρόκειτο να εφαρμόσουν αυτή τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών μεταχειρισμένων ρούχων τελικά αποφάσισαν να μην υπάρξει αυτή η απαγόρευση δείχνει ότι συνεκτίμησαν τα υπέρ κατά. Έκαναν τη δική τους ανάλυση Και αυτά έχω να σας πω να έχετε περαιτέρω ερωτήσεις. Πρόεδρος. Έχουν πιο ισορροπημένη άποψη λέτε. Αλλά φοβούνται ίσως ε, τις επιπτώσεις ε, της ε, ε, απαγόρευσης αυτής πρόσβασης στην αγορά των ΗΠΑ. Πάντα υπάρχουν δύο όψεις σε κάθε νόμισμα πριν από χρόνια. Λέγαμε ότι να εισαγάγουμε επιδοτούμενα τρόφιμα στην Αφρική. Και όταν είχα πάει στην Κάνα διαπίστωσα ότι επειδή το επιδοτούμενο ρύζι από την Αμερική καταργήθηκε, σταμάτησε η παραγωγή ρυζιού επιτόπου. Και μάλιστα ε, οι άνθρωποι εκεί θεωρούσαν ότι το αμερικανικό ρύζι είναι καλύτερο το δικό του αυτό που παρήγαν εκείνοι. Κάπως παρόμοια δεν είναι η κατάσταση. Διότι ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά μεταχειρισμένα ρούχα που είναι πολύ φτηνά και τα οποία συλλέγονται παγκοσμίω. Τα συλλέγουμε και μετά κάτι πρέπει να τα κάνουμε. Τα στέλνουμε σαν αναπτυσσόμενε χώρε Διάφοροι, ε, τα περισσότερα από αυτά τα δίδουν ε, ως πράξη φιλανθρωπίας ε, οι δικοί μας πολίτες. Δεν εξετάζεται λοιπόν η κατάσταση της επιπτώσης, των επιπτώσεων στην αγορά, λέτε. Δεν, δεν εξετάσατε τι ευρύτερες επιπτώσεις μπορεί να έχει στην ανάπτυξη των χωρών αυτών. Ναι, ανησυχείτε Τέλος πάντων, αλλά αν εξασχοληθούμε τώρα ιδιαίτερα με τα μεταχειρισμένα ρούχα, ξέρετε ότι εισάγονται σχεδόν τσάμπα. Πληρώνει κανείς δηλαδή μόνο για τη μεταφορά, γιατί συνήθως ε, τα ρούχα αυτά τα χαρίζουν οι πολίτες. Άρα, το φτωχότερο τμήμα του πληθυσμού που είναι σημαντικό ποσοστό σε αυτές τις χώρες. Σχεδόν 40% σε αυτές τις χώρες. Μπορεί να επωφεληθεί από αυτά τα ρούχα. Μπορεί να τα φορέσει. Είναι πολύ φτηνά. Δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν ούτε καν ε, τα κινέζικα εισαγόμενα ρούχα, τα οποία μαζικά εισάγονται στην Ανατολική Αφρική και εκπροσωπούν ένα μεγάλο τμήμα των εισαγωγών τους κλώστο εφαντουργικών και ρούχων. Άρα πρέπει να το δούμε και από τις δύο πλευρές. Αλλά μέχρι στιγμής θεωρούμε ότι το όφελος για τους πολίτες της περιοχής της Ανατολικής Αφρικής είναι σημαντικό και δεν θίγει τον κλάδο τοπικά, ο οποίος οπωσδήποτε πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστικός ιδιαίτερα για να μπορέσει να κάνει εξαγωγές προς τις ε, Ηνωμένες Πολιτείες και την Ένωση αλλά και για να μπορέσει να πουλήσει στους ε, ευπορότερους κατοίκους της περιοχής. Αλλά αυτά, πρόεδρος, πρέπει να το κοιτάξουμε περισσότερο. Γιατί, ξέρετε, αυτοί που κάνουν αυτές τις εξαγωγές δεν είναι φιλανθρωπικές οργανώσεις τελικά είναι ε, επιχειρήσεις. Και αυτοί έπεισαν ε, την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αναστείλει την πρόσβαση στις αγορές των ΗΠΑ σε αυτές τις χώρες. Πρέπει να δούμε λοιπόν τις αναπτυξιακές πλευρές. Αλλά πάση πρέπει να τα εξετάσουμε περισσότερο. Αλλά δεν είναι απλώς ε, ένα θέμα εμπορικών συναλλαγών. Γιατί οι χώρες της Ανατολικής Αφρικής θεώρησαν ότι ήταν αρκετά σημαντικό το θέμα για να αποφασίσουν να το απαγορεύσουν και τελικά υποχώρησαν λόγω των απειλών που υπέστησαν. Λοιπόν, τώρα. Υπάρχει εκπρόσωπος από την ε, Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Έχει έρθει. Α, χαίρετε, ευχαριστούμε. Ωραία, ερώτηση του κυρίου Γκεραέρο. Για τη διάσκεψη για τη Συρία που γίνεται, τι υποσχέσεις είχαν γίνει. Οι υποσχέσεις του 2017 όντως ε, υλοποιήθηκαν Έχετε την ερώτηση μπροστά σα, Παρακαλώ, κύριοι της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ, μήπως μπορείτε να μας πείτε το όνομά σας. Μαρτίν Αγγιλαντούτσι. Ασχολούμαι με το θέμα της Συρία στη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Συγγνώμη που άρχισα. Θα επιχειρήσω να απαντήσω στην ερώτησή σας. για τη χρηματοδότηση που αποφασίστηκε στην διάσκεψη Βρυξέλλες 1 από τα Ηνωμένα Έθνη και τα κράτη-μέλη. Η διάσκεψη αυτή έγινε στις 4 και 5 Απριλίου του 2017. Οι διεθνής κοινότητα και κυβερνήσει κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής προσφύγων τόνισαν τη δέσμευσή τους να βοηθήσουν τα εκατομμύρια των προσφύγων. Οι ενωσιακοί θεσμοί ε, υποσχέθηκαν 1,27 δις για το 2017 και η συνολική συμβολή των ενωσιακών θεσμών ήταν 1,42. Είναι 112% των ε, υποσχέσεών μας. Δηλαδή συνολικά τα κράτη-μέλη και η Ένωση υποσχέθηκαν 4,5 δις, που είναι 120% των υποσχέσεων που έγιναν στη διάσκεψη. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνεισφορές της Ένωσης και των κρατών μελών, δημοσιεύθηκε πρόσφατα μία έκθεση. Είναι διαθέσιμη στο site του Συμβουλίου. Ελπίζω να πάτε στην ερώτησή σας. Ενρίκε, θέλεις να ρωτήσεις τίποτα περαιτέρω. Καταρχάς ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ικανοποιητικό είναι ότι η συμβολή της Ένωσης ήταν πάντο, πάντα τελικά 100%, πάνω από 100% από όσα είχαν υποσχεθεί στην πρώτη διάσκεψη. Αυτό είναι θετικό. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όλοι μας. Αλλά το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης σε σχέση με τις ανάγκες Τη Συρία εξακολουθεί να υπάρχει. Παρά τη συμβολή τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Χθε στη διάσκεψή μας ήρθε ο αναπληρωτή γραμματέας της ΟΤΣΑ και μας είπαν ότι εκεί χρειάζονται περίπου 8 δις δολάρια για να καλύψουν τις ανάγκες των γειτονικών χωρών Λίβανος, Ιορδανία και Τουρκία. Τις ανάγκες που προκύπτουν από την κρίση στη Συρία δηλαδή. Οπότε, ικανοποίηση από τη μια γιατί τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας, μάλιστα υπερ τηρήσαμε τα υποσχεθέντα. Αλλά οι ανάγκες υπογραμμίζω ότι εξακολουθούν να είναι τεράστιες. Και κάτι ακόμη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε, θα είμαι ευγενικό. Γιατί εγώ είμαι από του πιο ευγενικού ευρωβουλευτέ σε αυτήν την επιτροπή. Αλλά θα πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μας αρέσει πολύ στο κοινοβούλιο να μας λένε πηγαίνετε να διαβάσετε στη σελίδα μας, στην ιστοσελίδα μας. Εμείς είμαστε το κοινοβούλιο που ελέγχει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε εκπρόσωποι των πολιτών που ελέγχουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι η κυβέρνηση της Ένωσης. Πολύ καλύτερο θα ήταν να μας δώσετε λίγη πληροφόρηση παρά να μου πείτε ότι αν θέλω περισσότερη πληροφόρηση να πάω στο ίντερνετ και να δω τι λέει στη σελίδα του Συμβουλίου. Και νομίζω ότι, νομίζω ότι αυτή είναι μια άποψη που βρίσκει σύμφωνα όλα τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης. Πρόεδρος, στο μέλλον να μας φαίνεται αυτά τα κείμενα. Γιατί πρέπει να μπορούμε να δούμε τι μας λέτε. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε πιέζοντας τις κυβερνήσεις μας εάν δεν πληρώνουν όσα υποσχέθηκαν. Και έχω μια συμπληρωματική ερώτηση. Εγώ και ο Νόρμπερτ Μόλις συναντηθήκαμε με συναδέλφους που ασχολούνται με την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων που ήρθαν σήμερα εδώ γιατί έγιναν δεσμεύσεις και υποσχέσεις στη διάσκεψη για τη Συρία το 16 και το 17 ότι όλα τα παιδιά από τη Συρία στην Τουρκία, το Λίβανο και την Ορδανία θα είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Θα πήγαιναν σχολείο. Και δεν ισχύει αυτό. Πολλές χιλιάδες παιδιών ακόμη δεν, μπορούν, δεν έχουν σχολείο να πάνε. Ωραία. Καλό είναι να υπόσχεστε ποσά. Αλλά υπέθετα ότι στα πλαίσια αυτά ένα συγκεκριμένο ποσό θα πήγαινε στην εκπαίδευση. Δηλαδή έχουμε μια συγκεκριμένη αναλυτική πληροφόρηση για το τι δαπανάτε γιατί. Γιατί δεν έχουμε τηρήσει την υπόσχεσή μας για το θέμα της εκπαίδευσης και είδα και κάποια στιγμιότυπα από τη διάσκεψη το 16 στο Λονδίνο και ο Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, τον David Κάμερον, πριν από την καταστροφική του απόφαση να κάνει δημοψήφισμα, είπε ότι όλα αυτά θα έχουν γίνει μέχρι τον Σεπτέμβριο. Και πριν από ένα χρόνο, νομίζω τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε υποθεί ότι όλα τα παιδιά θα μπορούσαν να πάνε σχολείο. Και εδώ είμαστε ακόμη δεν έχει γίνει. Δεν θέλουμε μόνο λοιπόν γενικά ποσά, αλλά πώ ξοδεύονται τηρούνται οι προτεραιότητές μας στι δαπάνε. Μπορείτε να μας πείτε τίποτα γι' αυτό. Ευχαριστώ. Να προσπαθήσω να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση για την αναγνώριση του κενού παρά τα θετικά στοιχεία που μόλις σας δώσαμε. Η Κομισιόν ε, το γνωρίζει αυτό πολύ καλά και προσπαθεί να φέρει περισσότερη χρηματοδότηση και να ε, διευρύνει και τον αριθμό των δωρητών. Και επίσης ε, περιμένουμε να δούμε ε, μετά από την διάσκεψη για τη Συρία την επόμενη μέρα να μπορέσουμε να έχουμε επαφή με τους δωρητές. Ε, τα σημειώνω όλα αυτά και θα διαβιβάσω τα μηνύματά σας και βεβαίως για το τρίτο σημείο για τις υποδείξεις είπα και για την παιδεία. Η παιδεία παραμένει το μέσο κλειδί για τις ε, επεμβάσεις της ε, ε, Ένωσης στην περιοχή αλλά και στην Συρία. Μέσα στην DG έχουμε την το πρόγραμμα εφαρμογής της ανθρωπιστικής βοήθειας και έχουμε έτσι γνωμοδότηση και συγκεκριμένους ανθρωπιστικούς εταίρους και ε, από αυτές τις βάσεις και επί τη βάση των ε, αναγκών που υποβάλλονται ε, στους εταίρους μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να δούμε πού πηγαίνουν τα χρήματα ανά τομέα. Παιδεία λοιπόν είναι μια από τις προτεραιότητές μας ε, μέσα στη Συρία. Διάφοροι εταίροι εφαρμόζουν προγράμματα εκπαιδευτικά, επίσημη και ανεπίσημη εκπαίδευση σε ολόκληρη την περιοχή. Δεν υπάρχει κάποιο ποσοστό το οποίο είναι αφιερωμένο στην παιδεία. Ας πούμε έχουμε χίλια λεφτά, τόσα θα πάνε στο παιδεία, τόσα στο ένα, τόσα στο άλλο. Για να μπορούμε να δούμε με διαφάνεια πού πάνε τα χρήματα. Όχι, η δέσμευση μπορεί να είναι για συγκεκριμένε χώρε, αλλά όχι για συγκεκριμένο τομέα αυτή τη στιγμή. Ρίκε, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, επόμενο σημείο είναι το 22 για το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο. Από με την προ με την Επιτροπή Προπολογισμού και δεν μπορούν να είναι εδώ παρά στις 17.45, οπότε πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα. Αλλά πριν κάνουμε διάλειμμα να δούμε στα διάφορα αν έχουμε τίποτα, οπότε να το έχουμε αυτό διεκπαιρεώσει. 25, επόμενη συνεδρίαση, 16 Μαΐου, στις 9 μέχρι το 12.30 και το απόγευμα και 17 Μαΐου το πρωί. 17 και 45 θα ξαναρχίσουμε γιατί είναι από κοινού. Α, 17 και 35. Σε 10 λεπτά θα είναι εδώ η Επιτροπή Προπολογισμού. Αν μου επιτρέπετε, κάτι δεν πήγε καλά. Αλλά έχουμε προσθέσει και εμείς μία προφορική. Κάπου εξυφανιστεί. Γιατί αν δεν υπάρχει κανείς εδώ να την απαντήσει, δεν χρειάζεται να την θέσω. Τι αφορούσε. Αφορούσε ε, την χρηματοδότηση από το ODA. Και από ό,τι είχα καταλάβει από τη γραμματεία θα ήταν για σήμερα. Αν όχι, ε, τότε δεν ε, έχει νόημα να θέσω την ερώτηση. Όχι, ε, συγγνώμη, εγώ έχω μόνο δύο ερωτήσεις, δεν έχω τίποτα για στο φωτοσχέ για τρίτη ερώτηση. Συγγνώμη, Τζούντιθ, εσύ δεν άρχισε και διαρωτήθηκα τι, γιατί ήρθες, αναρωτήθηκα γιατί ήρθες, αλλά εντάξει, όχι, μάλλον λάθος. Είχαμε και ένα σωρό ψηφοφορίες το πρωί. Την επόμενη φορά λοιπόν θα το δούμε. Ε, θα έχεις προτεραιότητα. Θα είσαι η πρώτη ερώτηση για την επόμενη φορά. Να την κρατήσουμε για την επόμενη φορά. Εντάξει. Περιμένουμε λοιπόν 10 λεπτά για το συναδέλφο της Επιτροπής Προπολογισμού.